Dank. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους της ΑΦΕΤ που είχαν την υπομονή να παραμείνουν εδώ. Έχουμε και τους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης και Πολιτικών Ελευθεριών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. έχουν έρθει εδώ για την παρουσίαση. Έχουμε και την κυρία Βαλενσιάνο εδώ. Θα συμπροεδρεύσουμε. Τιμούμε με το βραβείο Ζαχάροφ αξιόλογες προσωπικότητες που πολλές φορές με κίνδυνο ζωής και ελευθερίας αγωνίστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται, θα σας θυμίσω, για την έναρξη της διαδικασίας για τους υποψηφίους. Θα ψηφίσουμε την προσεχή εβδομάδα στην Επιτροπή για να επιλέξουμε τους τρεις εκ των οποίων το Προεδρείο θα διαλέξει έναν για να παρουσιάσει στις 22 Οκτωβρίου. Έχουμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο του Προέδρου. Το βραβείο Ζαχάροφ είναι η πλέον ε, ορατή πτυχή τη δουλειά που κάνει το Κοινοβούλιο για την πραγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αλλά βέβαια δεν είναι η μόνη. Επίση, για να μην έχουμε παρεξηγήσει την Τρίτη, σα υπενθυμίζω ότι δεν πρόκειται να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Για έναν πολύ απλό λόγο. Εάν κάποιος λάβει πάρα πολύ λίγες ψήφους και αυτό καταστεί γνωστό δημόσια, πλήττεται η εικόνα το κύρος του και βέβαια δεν τον βοηθούμε καθόλου στη χώρα του εάν τυχόν έχει κίνδυνο διώξεων. Δεν ναι, σωστό λοιπόν αυτό. Παρακαλώ λοιπόν να μην μιλήσουμε για τα θέματα αυτά στα μέσα μαζική ενημέρωση. και επίση να μην δημοσιευθούν και τα, ε, τα αποτελέσματα για, ή τα στοιχεία ακόμα για τους τρεις πρώτους, να μην μαθευτούν τα τρία πρώτα ονόματα, ώστε να προχωρήσουμε κατά τρόπο απρόσκοπτο. Και συνήθως ξέρετε ότι μέχρι τώρα όποτε κάποιος ήταν πρώτος στη λίστα τη δική μας, ήταν και αυτός που τιμήθηκε εν τέλει από το Προεδρείο. Είναι αρκετά διαφανείς διαδικασίε εδώ. Ενώ στο βραβείο Νόμπελ κανείς δεν γνωρίζει πώς γίνονται οι επιλογές. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχουν γίνει συζητήσεις για ε, έλλειψη διαφάνειας και άλλα τέτοια. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυσικά το παίρνουμε υπόψη μας πάντα. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω το ρόλο στις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ το προσωπικό πάντως που με βοήθησε, που μου έγραψε ένα πολύ καλό κομμάτι εδώ. Και θα περάσουμε στους υποψηφίους. Οι ευρωβουλευτές όπως ξέρετε, παρουσιάζουν υποψηφίους. Τους υποψήφιους δηλαδή εδώ σήμερα 10 λεπτά για τον καθένα θα διαθέσουμε και 40 λεπτά συνολικά για την παρουσίαση των υποψηφίων. Αρχίζουμε με τη σειρά, την αλφαβητική, ελευθερία συνείδησης και έκφραση στην Τουρκία, κάνουν ντούνταρ, από την ΚΟΕ, τους Πράσινους και το LDD. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βερζιά πρώτα απ' όλα. Για τρία λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχετε δίκιο που επιμένετε για τη σημασία που έχει το βραβείο Ζαχάροφ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όντως, είναι πολύ σημαντικό και προς το εξωτερικό και χαίρομαι που φέτος μπορούμε να υποβάλουμε από κοινού τρεις πολιτικές ομάδες την υποψηφιότητα του Καντούνταρ που είναι ένα πραγματικό σύμβολο, σύμβολο για το τι τραβάνε οι δημοσιογράφοι στην Τουρκία, ε, σύμβολο των ε, συνεχιζόμενων και αυξανόμενων απειλών των οποίων είναι θύματα. Είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος, κάνει έρευνες, κάτι το οποίο ποτέ δεν ήταν εύκολο στην Τουρκία και εδώ και πολλά χρόνια τα πράγματα χειροτερεύουν. Ήδη το 2012 οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου όσον αφορά τους δημοσιογράφους και μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής ε, έντασης από το 2015 τουλάχιστον τα πράγματα κάθε άλλο παρά έχουν βελτιωθεί. Ο Τσεντουντάρ λοιπόν είναι ένας δημοσιογράφος από τα 18 του. Έχει δίπλωμα από το London School of Journalism δούλεψε στην Τουρκία, στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και συμμετείχε στην ε, παραγωγή πολλών ε, πολλών ε, ντοκιμαντέρ και το 2015 η Κουμχουριέτ δημοσίευσε κάποια έγγραφα τα οποία ενοχλούσαν την κυβέρνηση. Με έδειχνε δηλαδή φορτηγά τα οποία πηγαίναν όπλα προς τη Συρία. Υποτίθεται ότι μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και συνοδεύονταν από την MIT που είναι η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών. Στα σύνορα λοιπόν του σταμάτησαν οι ίδιοι Τούρκοι χωροφύλακες και αυτοί συνελήφθησαν επειδή είχαν αποκαλύψει κρατικά μυστικά. Τον Ιούνιο ο ίδιος ο Ερτοκάν υπέβαλε μήνυση κατά του Τσεντούνταρ λέγοντας ότι αυτός έπρεπε να πληρώσει την νύφη και μάλιστα ζήτησε και ισόβια φυλάκιση γι' αυτόν. Πρόεδρε, πρόεδρε, αν ε, δεν μιλούσατε πιο δυνατά από ό,τι μιλάω εγώ, θα ήταν καλό για να συνεχίσουμε τη συζήτηση εδώ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Βερζιά. Συνεχίζω λοιπόν. Στις 26 Νοεμβρίου που μας πέρασε, ο Τζάνα Τουντάρα ε, συνελήφθη και πέρασε 90 μέρες στη φυλακή. Τον Μάιο του 2016 γλίτωσε από δολοφονική απόπειρα μπροστά στο δικαστήριο ενώ πήγαινε σε μια συνέντευξη τύπου για να σχολιάσει την καταδίκη του. Μετά έγινε μια πραγματική απόπειρα πραξικοπήματο, το ξέρουμε όλοι, και η καταστολή επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο στην Τουρκία και η ελευθερία τύπου είναι καινή λέξη. Στις 26 Ιουλίου ε, διετάχθη να κλείσουν 45 εφημερίδες, 7 τηλεοπτικοί σταθμοί, υπηρεσίες τύπου, 15 περιοδικά κλπ. Έχουν ε, ακυρωθεί πάρα πολλές εντεύξεις τύπου και 200 τόσοι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, από τους οποίους οι μισοί εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή. Σε έκθεσή τους οι γιατροί χωρίς σύνορα λένε ότι πλήττεται η ελευθερία στην Τουρκία όσο ποτέ. Ο Δε Τσαντουντάρ έφυγε από την Τουρκία γιατί είπε ότι δεν εμπιστεύεται πια τη δικαιοσύνη της χώρας του. Η γυναίκα του όμως συνελήφθη. Το διαβατήριό της, ε, της το πήραν για να εκβιαστεί ο Τσαντουντάρ να επιστρέψει στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε συνάδελφοι γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αξίζει το βραβείο Ζαχάροφ γιατί ακριβώ συμβολίζει όλη αυτή την καταπίεση και την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Η ομάδα μου των Πρασίνων θέλει να προτείνει τον ε, κινηματογραφιστή και δημοσιογράφο Τσάντουν Ντάρ ε, για το βραβείο ε, ελεύθερης έκφρασης και σκέψης του βραβείου Ζαχάροφ. Εδώ και χρόνια αποδίδεται στους πλέον αξιοθαύμαστος υπερασπιστές της ελευθερίας το βραβείο αυτό και πιστεύουμε ότι ο Τσάντουν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία ε, των σύγχρονων ηρώων και μάλιστα στις πρώτες θέσεις. Είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα της τουρκικής δημοσιογραφίας. Είναι ένα ζών σύμβολο της ε, ελεύθερης ε, σκέψης και έκθεσης στη χώρα του. Τα τελευταία 35 χρόνια έχει αγωνιστεί παθιασμένα για την ελεύθερη και τον ελευθεροτυπία και την ελεύθερη έκφραση. Έχει αγωνιστεί για μη βίαιη μάλλον για ε, όλο ένα και κοντινότερη προσέγγιση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρξε πηγή έμπνευση για πολλούς από εμά στην Ευρώπη και στην Τουρκία το ίδιο. Επίσης, έχει συνηγορήσει ανοιχτά υπέρ της ειρήνης, της ε, δημοκρατικής επίλυσης και της ειρηνικής επίλυσης του κουρδικού ζητήματος. Το τελευταίο καιρό διώχθηκε βία και ε, από την κυβέρνησή του, γιατί αποκάλυψε κυβερνητικά μυστικά. Συνελήφθη, ε, κρατήθηκε στην απομόνωση και υπέστη σοβαρή και υπέστη μάλλον μια ε, βαριά ε, ποινή. Ε, μετά την αποτυχημένο απορριξικόπημα φέτος το καλοκαίρι χρειάστηκε να φύγει από τη χώρα του, να διαφύγει λόγω της αβεβαιότητας για τη σωματική του υγεία και του νομικού κενού καθώς και της αβεβαιότητας ε, με τα καθεπίγοντα μέτρα. κατασχέθηκε το διαβατήριό του εντωμεταξύ και η Τουρκία είναι μια από τους κοντενότερους γειτονές μας και εταίρους. Είναι επίσης υποψήφια για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λαοί της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν πάντοτε στενούς δεσμούς. Έχουμε δεσμούς μέσω του πολιτισμού, της ιστορίας, της οικονομίας και με πολλές προσωπικές ιστορίες. Ε, για την Συρία και πολλά άλλα ε, κομμάτια της γειτονιάς μας σίγουρα φλέγονται αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν και άλλες σχέσεις στο άμεσο περιβάλλον μας που είναι ίσω πιο σημαντικέ από τι σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, όμω βλέπουμε διαρκή υποβάθμιση της προστασίας ανθρωπινών δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. στη χώρα αυτή. Βλέπουμε διαρκώ να υπάρχουν εντάσεις στι σχέσει μα και στι πρωτεύουσε μα, οι ηγέτες μα και οι κρατικοί φορεί αρχίζουν να παραδίδουν τα όπλα για τι πιο βασικέ αξίε και αρχές στο όνομα μια κοντόφθαλμη και ε, πολιτική για την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Η Ευρώπη στρέφει τα νότα τη ε, και παραμελεί την Τουρκία. Ενώ αυτοί που προασπίζονται τη δημοκρατία κατά του απολυταρχισμού αυτοί που δεν θέλουν να ξαναρχίσει ο πόλεμος και ο ανθρώπινος πόνος σε αυτές τις περιοχές δεν προστατεύονται. Εάν αποδώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ 2016 στον ε, Τζαν Ντουντάρ, το κοινοβούλιο ουσιαστικά αποτεί φοροτιμή στον εαυτό του, διότι θυμίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ότι η πολυφωνική και δημοκρατική Τουρκία είναι κάτι το οποίο επιθυμούμε. Εάν το αποδώσουμε αυτό το βραβείο, ε, το Ευρωκοινοβούλιο θα αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα από τι Βρυξέλλε, ότι η κατάσταση στην Τουρκία έχει σημασία. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σκοπεύει και δεν πρόκειται να καταλήψει τους υπερασπιστές μιας ζωντανής ε, εύρος της Τουρκίας την οποία ε, όλοι αγαπάμε και θέλουμε να είναι καλά σήμερα. Η ελευθερία και η ζωή του Τσάν Τουντάρα απειλούνται ε, επειδή δημοσίευσε συγκεκριμένα άρθρα στον τύπο. Πρέπει να το στηρίξουμε και όλες τις ελεύθερες φωνές της Τουρκίας. Γι' αυτό τον προτείνουμε ως υποψήφιο για το βραβείο Ζαχάρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μένα είναι τιμή και μεγάλη χαρά να μπορώ εξ ονόματος της ομάδας μου αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων από κοινού να υποβάλω την υποψηφιότητα του Τσάν Ντουντάρη για το βραβείο Ζαχάροφ. Το βραβείο Ζαχάροφ, όπω υπόθηκε προηγουμένω, είναι ένα βραβείο που αποδίδεται στην ελευθερία τη σκέψη. Εάν δούμε τη διαδρομή του τα τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι η Τουρκία έχει επίσημο ε, ε, καθεστώ υποψήφιο χώρα από τα 99, 17 χρόνια τώρα. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι η ελευθερία τη έκφραση και η ελευθεροτυπία, ε, η ελεύθερη έκφραση είναι στα θεμέλια του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώ ένα γεωγραφικό χώρο ή ένα πολιτικό εγχείρημα. Είναι μια ιδέα που βασίζεται στο γεγονό ότι μπορεί να υπάρξουν διαφορετικέ αποκρίσει στην ίδια ερώτηση. Οπότε θα πρέπει να δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ε, απομακρύνεται από αυτό το ιδεώδε ένα και περισσότερο το σημερινό τουρκικό κράτο. Ο Τζαν Ντουντάρ θα πρέπει να λάβει αυτό το βραβείο, διότι αυτοί οι αρχέ ε, είναι κάτι που προασπίστηκε ε, όλη του τη ζωή και πλήρωσε και το ανάλογο τίμημα, χειρότερο από τον ε, θάνατο, την εξορία, μακριά από του δικού του και τη χώρα του. Εάν αποδώσουμε το βραβείο αυτό στον Τζαν Ντουντάρ, το αποδίδουμε σε όλου αυτού που είχαν την ίδια τόλμη που το κάνουν αυτό συχνά και που αντιμετώπισαν δυσκολίε και δεν ανταμείφθηκαν ποτέ. Μόνο και μόνο γιατί εκφράστηκαν ελεύθερα. Ε, ύψωσαν τη φωνή του, απέναντι σε μια πολιταρχική εξουσία και ενημέρωσαν ε, τον υπόλοιπο πληθυσμό για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης. Ε, αυτές που ε, τους φέρνουν σε δύσκολη θέση, αυτές που είναι επικίνδυνες, όπως με τις αποκαλύψεις του Τσάντουν Τάρκετ της εφημερίδας τα τελευταία χρόνια. Στην Τουρκία φυλακίστηκαν 120 δημοσιογράφοι τα τελευταία χρόνια και πάνω από 100 ε, πρατήρια νομιστή που ε, έχουν κλείσει. Η χώρα είναι στην 150η ε, θέση από τις 180 χώρες ως προς την ελευθερία έκφραση του τύπου. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων η Τουρκία. Είναι μια χώρα, όπως υποθυμώ και προηγουμένως, για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμως. Ε, το θέμα αυτή τη υποψηφιότητα είναι θέμα χρόνου. Έχουμε ακόμη το περιθώριο του χρόνου να ε, κάνουμε κάτι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Μια στιγμή ουσιώδη. Θα μπορούσαμε να θυμίσουμε ότι η χώρα αυτή απομακρύνεται μοιραία, όχι μόνο από οποιαδήποτε προοπτική εισόδου στην ε, Ένωση, αλλά και από οποιαδήποτε σύγκληση προ τι αξίε μα. Δεν πρέπει να, έχουμε, να φοβόμαστε να καταγγείλουμε αυτή την απόκληση, να θυμίσουμε ότι η Τουρκία ασφάλει, ότι το επάγγελμα των δημοσιογράφων ε, πρέπει να είναι ελεύθερο να εκφραστεί για να εκφράζει τις αισθήσει και τι ανάγκε των ίδιων των πολιτών. Οι πολιτικέ σκοπιμότητες δεν μπορεί να προηγούνται σε σχέση με τι κατάφορε παραβιάσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα ήμασταν συνένοχοι αν δεν το αποκαλύπταμε, αν δεν το καταγγείλαμε. Η ψήφη μα, λοιπόν υπέρ του Τσαντουντάρ δεν είναι ψήφο κατά τη Τουρκία, είναι στήριξη τη κοινωνία των πολιτών τη χώρα αυτή. Είναι μια ελπίδα για το μέλλον. Εάν καταδικάστηκε σε εξορία ο Τσάντουν Ταρ ε, εμεί θέλουμε να εμποδίσουμε να καταδικαστεί ο ολόκληρο τοπικό λαό να ζει σε ένα δημοκρατικό κράτο και όχι μόνο όνομα. Να μην εξοριστεί από το κράτο δικαίου. Ο Ζαχάροφ έλεγε ότι μέχρι μια χώρα να αποκτήσει ελευθερία για του πολίτε τη στην πληροφόρηση και με ανεξάρτητο τύπο, τότε δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για την κοινή γνώμη ώστε να ελέγχει την συμπεριφορά τη κυβέρνηση. Σήμερα θέλω να σα το θυμίσω και να το θυμόμαστε πάντοτε διαρκώ όλοι μαζί και Γι' αυτό να ψηφίσουμε υπέρ της υποψηφιότητας. Ευχαριστώ. Μουσταφά Τζέμιλεφ. Uh, uh, Πρόταση του ΕΛΚ και του ECR. Σάριος Βόλφσκι. 1 και 45. Είναι ένας μοναχικός αγωνιστής κατά της ε, δικτατορίας. Μα είναι και η ίδια η ουσία του γραφείου Ζαχάροφ. Δεν υπάρχει άλλος που να είναι πιο κοντά στο μοντέλο αυτό που έχουμε για το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι αυτός που συνεχίζει χωρίς βία να αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, κατά της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσίας έχοντας θέσει και κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, όπως αναφέρουμε και στο φυλαδιό μας. Ε, στην ε, Κρυμαία, γεννητική έφυγε, έζησε σε εξορία και διαμαρτυρήθηκε ήδη για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στη Τσεχοσλοβακία και πέρασε πολύ καιρό στη φυλακή. Σήμερα συνεχίζει τον αγώνα του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, στην Κρυμαία, και κυρίως για τους δικούς του, του στάταρους της ε, Κρυμαίας. Από το 1944, όπου τον έδιωξαν από την ε, Κρυμαία και 70 χρόνια μετά ε, πάλι τον έδιωξαν από την Κρυμαία. Την πρώτη φορά η Σοβιετική Ένωση, τη δεύτερη φορά η Ρωσία. Συνεχίζει λοιπόν να δίνει αγώνα για την ελευθερία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και η ομάδα μας προτείνω σε υποψήφιο τον Μουσταφά Τζεμιλέφ για το βραβείο Σαχάροφ και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε και ένα μικρό βίντεο να σας παρουσιάσουμε. Δεν ξέρω, ο τεχνικός θα έπρεπε να είναι έτοιμο για το βίντεο αυτό, αλλά δεν ξέρω. Είναι. Πού είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μουσταφά Τζεμιλέ είναι εξέχουσα προσωπικότητα ο οποίος ασχολείται με τα δικαιώματα των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και των μειονοτήτων. Από το 1996 που συνελήφθη, πέρασε 15 χρόνια στις φυλακές. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ήταν από αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν για την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία και μετά κατά τη διάρκεια της άνοιξης της Πράγας αγωνίστηκε επίσης. Οπότε είναι και ένας από τους πρώτους που στήριξαν και το βραβείο μας. Τώρα, για άλλη μια φορά, τον έδιωξαν από τη χώρα που γεννήθηκε, από την Κρυμαία, από τους ε, Ρώσους. Είχε συμβεί ήδη αυτό όταν ήταν 6 μηνών από την τότε Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα για κάποιον ο οποίος ε, υψώνει τη φωνή του για να καταγγείλει τέτοιες παραβιάσεις. Για κάποιον που στηρίζει τα δικαιώματα των ε, Ουκρανών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε με τον, ε, με την υποψηφιότητά του αυτή και να του δώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πολωνός συνάδελφος βρίσκεται στην Ορθανία σήμερα. Από εκείνον ήρθε αρχικά η προϋποψηφιότητα. Παρουσιάζω λοιπόν τον υποψηφία εκ μέρους του. Πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε πολλού σοβαρού υποψηφίου φέτο και παρακολουθώ όλε αυτέ τι εξελίξει τα τελευταία χρόνια, τις υποψηφιότητες, όμως ο κ. Ντεμιλεύ είναι ιδανικό υποψήφιο, διότι όπως είπε ο Ζαχάροφ, είναι πρώην ε, σοβιετικό αντιφρονούντα ε, αντιφρονούντας και έχει προασπιστεί τον αντιφρονών και έχει ένα ε, μακρό, μακρόχρονο βιογραφικό για την ε, καταπολέμηση για την διαφωνία του με το κομμουνιστικό καθεστώς στην εποχή του Στάλιν απελάθη, όταν ήταν ακόμα εξάχρον, εξάμεινο μωρό, και επιστρέψει στην Σοβιετική Ένωση το 1968 ήταν από του πρωτηγέτε για την προστασία των δικαιωμάτων τη Σοβιετική Ένωση και με την εγκρίση τη πέρασε 16 χρόνια στη φυλακή στη Σοβιετική Ένωση, ένα χρόνο απεργία πείνα σχεδόν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά την προσάρτηση τη Κρυμαία από τη Ρωσία. εξέφρασε την καταδίκη του κατά τη προσάρτηση και βεβαίω το απογραφική είσοδο στην πατρίδα του, την αιστεία των Τατάρων. Εδώ η ε, Ρωσία εμποδίζει την ε, πορεία της Ουκρανίας προς τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και βεβαίως ο κ. Ντεμιλέφ εκφράζεται κατά της πίεσης αυτής. Δέχεται τις ίδιες πιέσεις ακριβώς από το κράτος που διαδέχτηκε την Σοβιετική Ένωση, την Ρωσική Ομοσπονδία και ο ίδιο και ο λαό του. Έχει αγωνιστεί στη δικαιοσύνη και 17 χρόνια μετά την απέλαση 25 χρόνια μετά την επιστροφή του στη χώρα του, εκπροσωπεί ε, την ηθική και πνευματική ηγεσία του διεθνού κινήματο των Τατάρων ε, για την εξαρτησία του. Θέλει ε, να παραμείνει η Κρυμαία στην. Ουκρανία και αγωνίζεται για τα δικαιώματα του λαού του. Μετά τις απειλές ε, από τη Ρωσία προς την Ανατολική Ευρώπη και τις απειλές κυβερνητικού πολέμου με την προπαγάνδα και την ε, μηχανή προπαγάνδας που κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζω ότι το, το βραβείο Ζαχάρα πρέπει να αποδοθεί σε αυτόν τον, ε, τον αντιφρονούντα, γιατί ακριβώς Τάταροι είναι σύμβολο για, τις, ε, για τους λαούς των οποίων τα εδάφη δέχονται εισβολή και ζουν σε κατοχή. Έχω συναντήσει τον κύριο Τζεμιλέφ αρκετές φορές, όπως πολλοί από τους συναδέλφους στο Ευρωκοινοβούλιο και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι, ένα πολύ, πολύ, είναι ένας πολύ σοβαρός υποψήφιος για τον Ροδίο Ζαχαρό.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 Συνεχίζουμε. Ο κύριος Μπροκ θα φύγει σε λίγα λεπτά. Οι επόμενες υποψηφιότητες στη φετινή εκλογή είναι η Νάντια Μουράντα και η Λαμίγια Αλή Μπασάρ που τις προτείνουν οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι, το ΑΛΔΕ. Οπότε ένας από κάθε μία από αυτές τις δύο πολιτικές ομάδες θα μας τις παρουσιάσει. Για πέντε λεπτά πρώτα ο συνάδελφος Βαντεχόλσελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αποφάσισε σήμερα για φέτος να παρουσιάσει τις δύο αυτές υποψηφιότητες των δύο πρώην θυμάτων σεξουαλικών σκλάβων των, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους. Για να τιμήσει το θάρρος τους, να ξεφύγουν από την εξουσία των, του, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους και για το θάρρος που έδειξαν προσπαθώντας να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Οι Γεζιδίτες ζουν στα βόρεια του Ιράκ, είναι τώρα πολλοί από αυτούς ήδη στην Ευρώπη. Η οργάνωση που ονομάζεται Ισλαμικό κράτος έχει αναπτύξει τη θεολογία των βιασμών που συστηματικά εφαρμόστηκε στις γυναίκες και τα κορίτσια που απήγαγαν από την κοινότητα των γεζιδιτών όταν καταλάμβανε το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος στα ε, εδάφη τους ε, και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούσε ως ε, σεξουαλικές σκλάβες αυτό από τον Αύριο του 2015 όπου, στα, όπου έφτασε το Ισλαμικό κράτος στο βορειοδυτικό Ιράκ στα σύνορα με τη Συρία πάνω από 6.000 γυναίκες έχουν απαχθεί γυναίκες και κορίτσια απάγονται, συλλαμβάνονται, μεταφέρονται σε άλλες περιοχές του Ιράκ και της Συρίας για να χρησιμοποιηθούν ως σεξουαλικές σκλάβες, εγκλήματα αδιανόητα, 3.000 γυναίκες και κορίτσια θα μπορούσαν να απελευθερ... μπόρεσαν να απελευθερωθούν ε, ή να δραπετεύσουν από την κράτηση αυτή. Με την τίμηση των δύο αυτών υποψηφίων λοιπόν θέλουμε να τιμήσουμε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που είναι θύματα των συγκρούσεων, των εθνοτικών ε, ε, συγκρούσεων, της γυναικοκτονίας. Το Ισλαμικό κράτος στόχευσε κορίτσια και γυναίκες και χρησιμοποίησε με τον τρόπο αυτό το συστηματικό βιασμό για εθνοτικές καθάρσεις. Τακτική που είδαμε και στη Βοσνία και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στην Αφρική. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται η ιστορία. Απλώς οι δράστες είναι διαφορετικοί. Πρόκειται λοιπόν για ένα μήνυμα σημαντικό για τους εγκληματίες αυτούς. Πρόκειται και για ένα μήνυμα για την κοινότητα των Γεζιδιτών, που πάντοτε είναι η λησμονισμένη κοινότητα. Τώρα που βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της ιστορίας, το πιο δύσκολο σημείο της ιστορίας της, να τη δείξουμε ότι δεν την έχουμε ξεχάσει. Και επίσης θα πρόκειται και για τους πρώτους υποψηφίους από το Ιράκ. Ελπίζω να μας υποστηρίξουν στη διπλή αυτή υποψηφιότητα και οι άλλες ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπεθέρα έχει τώρα το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω και δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματα του συναδέρφου. Γιατί και εμείς υποστηρίζουμε την ίδια υποψηφιότητα. Πρόκειται για δύο νέες γυναίκες, θύματα και φοβερά θαραλές. Αποφάσισαν να μην είναι πια θύματα, αποφάσισαν ότι υπέφεραν ότι ήταν θύματα και όντω ήταν όλων των βιαίων πράξεων και παραβιάσεων και των δικαιωμάτων τους κτλ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση για αυτή την υποψηφιότητα. Ε, με την ε, Νάντια Μουράντ είχαμε περισσότερες επαφές, ε, την Λαμίγια την γνωρίσαμε αργότερα. Ελπίζω να τις στηρίξετε. Ήδη από τον Φεβρουάριο γνωριστήκαμε και εδώ στο Στρασβούργο ήρθε η Νάντια και αξίζει τον κόπο να ακούσουμε από τα δικά τους τα χείλη όχι μόνο το τι υπέφεραν αλλά και την εμπιστοσύνη που έχουν στη δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αυτή ακριβώ και είναι η βάση της υποψηφιότητας που προτείνουμε οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι. Θέλω να επιμείνω επίσης ότι δεν προτείναμε την Άντια Μουράντ μόνο επειδή είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα της ΔΑΕΣ ή επειδή ε, σκοτώσανε ολόκληρη την οικογένειά της ή τις βασανίσανε κτλ. Όχι, αλλά γιατί ακριβώς αποφασίσαν να μην είναι πια θύματα. Γιατί αποφασίσαν να κάνουν την αλλαγή και να αντιμετωπίσουν τον φανατισμό και να βοηθήσουν στη διαδικασία που θα οδηγήσει σε δικαίωση όταν οι υπεύθυνοι πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο. Νομίζω ότι στην Άντια, στη Λαμίγια και σε όλα τα θύματα πρέπει να δώσουμε το βραβείο Ζαχάροφ για να τους δώσουμε βοήθεια να μπορέσουν να ελευθερώσουν τις 3.000 και γυναίκες και κορίτσια που εξακολουθούν να είναι στη σκλαβιά και οι υπεύθυνοι να πάνε στο δικαστήριο. Το βραβείο αυτό ο Ζαχάροφ λοιπόν θα αποτελέσει μια αναγνώριση θα τις προβάλλει, αλλά πρόκειται και για πόρους που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι, υποστηρίζοντας κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη δράση. Θα επαναλάβω εδώ και τα λόγια της ε, Νάντια που τα γνωρίζετε μάλλον, γιατί έχει εδώ και πάνω από ένα χρόνο που έχει γυρίσει τον κόσμο ολόκληρο, έχει πάει στα Ηνωμένα Έθνη και έχει μιλήσει εκεί πριν από δύο ε, εβδομάδες μάλιστα την ορίσανε πρέσβυρα καλής θελήσεως. Έχει έρθει και εδώ με τον πρόεδρό μου τον κύριο Σούλτς, έχει συναντηθεί προσωπικά, έχει πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Παντού έχει πάει. Με έχει μιλήσει με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αυτό όμως που θα ήθελα εγώ να επαναλάβω εδώ είναι μια φράση της Νάντιας που νομίζω ότι καθορίζει τι σημαίνει αυτή η υποψηφιότητα. Είπε ότι η πήρε την οικογένειά μου, το μέλλον μου, τη ζωή μου. Αλλά μου μένει η καρδιά μου και πάντα θα την έχω, πάντα την είχα, όπω επίση και την πίστη μου στη δικαιοσύνη. Και όλε οι γυναίκε και τα κορίτσια που βρίσκονται στα χέρια των τρομοκρατών πρέπει να ξέρουν ότι η δικαιοσύνη είναι μαζί του, είναι στο πλευρό του. Αυτά είναι τα λόγια τη υποψήφια αυτή και αυτό ακριβώ είναι και το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι μια υποψηφιότητα δηλαδή η οποία ερμηνεύει όσο γίνεται καλύτερα και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις αξίες του βραβείου Ζαχάροφ που είναι η ελευθερία έκφρασης, η προστασία των μειονοτήτων, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, δημοκρατία, κράτος δικαίου. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι κατά μια τέτοια υποψηφιότητα γιατί πρόκειται για γενικές αξίες. Θα σας το πω και πάλι, πρόκειται για δύο αξιοθαύμαστες γυναίκες, νέες με φοβερό θάρρος που όσο γίνεται καλύτερα αντικατοπτρίζουν το ίδιο το πνεύμα του βραβείου Σαχάροφ. Για να τελειώσω λοιπόν θέλω να ε, πω και πόσο ευχαριστώ την Γερμανία που τις έχει υποδεχτεί. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος και αποτελεί ένα παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό εδώ. Οποιοδήποτε Γερμανός θα έπρεπε να νιώσει πολύ υπερήφανος ψηφίζοντας για την άδεια. Για διαδικαστικούς λόγους πρέπει να σας πω ότι δύο αυτές οι υποψηφιότητες τελικά ενώνονται της Νάντια και της Λαμίγια δηλαδή γιατί πρόκειται για τις ίδιες αξίες. Είναι καθαρά τεχνικό, οπότε εμεί συμφωνούμε με τι δύο αυτέ υποψηφιότητε και έτσι δεν έχουμε χωριστή υποψηφιότητα εμεί για την Νάντια Μουράντα, Αλλά η Νάντια Μουράντα με την Λαμίγια Άγιε Πασάρ πάνε μαζί και είναι υποψηφιότητε που προτείνουμε μαζί οι σοσιαλιστέ και εμεί. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπεθέρα. Κύριε Πρέντα, και εσείς έχετε να παρουσιάσετε υποψήφιο. Η κυρία Μπεθέρα τα εξήγησε. Θέλετε να τα επαναλάβετε κι εσείς. Μα εδώ φαίνεται, μα μόλις το εξήγησε η κυρία Μπεθέρα. Μόλις το εξήγησε. Μπορείτε κυρία Μπεθέρα να το εξηγήσετε και πάλι στα αγγλικά. Εγώ είμαι σίγουρη, λέει η κυρία Μπεθέρα, ότι η διερμηνία ήταν απόλυτα σωστή. Ίσως δεν το παρακολουθήσατε καλά. Λέω ότι υπάρχει μία υποψηφιότητα. Νάντια Μιράντ και η Λαμίγια Άγιε Μπασάρ αποτελούν μία υποψηφιότητα. Μα ακριβώς αυτό σας είπα, ότι για τεχνικούς λόγους, για διοικητικούς λόγους, ενώθηκαν οι δύο υποψηφιότητες. Προηγουμένως υπήρχε υποψηφιότητα της Νάντια Μουράτ που ήταν δικιά μας και η υποψηφιότητα της Νάντια Μουράτ και της Λαμίγια Άγιε Μπάσαρ που ήταν η πρόταση των σοσιαλιστών. Τώρα αυτά τα δύο ενώθηκαν. Δεν θα χωρίσουμε, δηλαδή δεν θα πούμε ότι είναι δύο υποψηφιότητε, είναι μία γιατί πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα. Την Άντια Μουράτ και τη Λαμίγια Άγιε Μπασάρ. Ο κύριο Πρέντα εκτό μικροφώνου είναι μία υποψηφιότητα που προτείνουν δύο πολιτικές ομάδες, οι σοσιαλιστές και η Άλντε. Πριν η Άλντε είχε προτείνει μόνο την Άντια Μουράτ. Τώρα προτείνουμε και εμείς και τις δύο. Οπότε είναι μία υποψηφιότητα τα δύο αυτά πρόσωπα από δύο πολιτικές ομάδες. Κοινή υποψηφιότητα. Η διαφορά είναι ότι η Άλντε προηγουμένως πρότεινε μόνο την Άντια, ενώ οι σοσιαλιστές πρότειναν δύο κυρίες. Λοιπόν, εμείς δεχόμαστε να υπάρξει κοινή υποψηφιότητα από τις δύο πολιτικές ομάδες και για τις δύο κυρίες. Οπότε εμείς αποσύρουμε τη δικιά μας υποψηφιότητα για τη μία κυρία και δεχόμαστε εκείνη των σοσιαλιστών και την υποστηρίζουμε για τις δύο κυρίες. Πρόεδρος, ό,τι θέλουμε μπορούμε να συνδυάσουμε είναι απλό. Οι σοσιαλιστές υπέβαλαν υποψηφιότητα για δύο γυναίκες και ζητήτες. Οι φιλελεύθεροι πρότειναν μία από τις δύο κυρίες. Οι φιλελεύθεροι τώρα συμφωνούν να υπάρχει υποψηφιότητα για δύο κυρίες και όχι για μία. Οπότε υποστηρίζουν την υποψηφιότητα αυτή για τις δύο κυρίες και οι δύο πολιτικές ομάδες. Είναι μία υποψηφιότητα για δύο γυναίκες που υποστηρίζουν δύο πολιτικές ομάδες. Και περνάμε στις επόμενες υποψιότητες. Ο επόμενος, Ήλαν Τότι. Ο συνάδελφός μας, ο Ήλαν Κιντσιούκ, ε, την προτείνεται υποψηφιότητα αυτή, μαζί με 42 άλλους ευρωβουλευτές. Έχουμε και ένα βίντεο και θα ακούσουμε και τον ε, συνάδελφο. Ναι. Πρόεδρε, έχω τη χαρά και τιμή να παρουσιάσω την υποψηφιότητα του Ιραντόχτη για, την, ε, για το βραβείο Ζαχάροφ του 2016. Μπορώ, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής Λαντόχτη λοιπόν είναι καθηγητής οικονομικών στο Χιντζάγκ ε, της ε, Κίνας και στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, γεννήθηκε το 1969, στο Χιντζάν και για 20 χρόνια ε, ειρηνικά προήγε τον διάλογο μεταξύ των Ούντου και των, ε, των Ουιγούρων και των Κινέζων ε, και προήγαγε ισότιμα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και ε, πολιτικά δικαιώματα. Τα 11 εκατομμύρια των Οιγούρων ζουν στη βορειοδυτική Κίνα. δεν έχουν απολαύσει τη, τα, τους καρπούς της ανοικονομικής ανάπτυξης της Κίνας των τελευταίων ετών. Αντιθέτω, έχουν πέσει θύματα κατασταλτικών πολιτικών και ανοιχτό τη ε, διακριτική μεταχείρισης και προφανώς διακριτική μεταχείριση ε, από τις κινεζικέ αρχές. Ο Ιλάν Τόχτη λοιπόν καταδικάστηκε σε φυλάκιση για απόσχηση. Κατηγορία γελία για, για άνθρωπο ο οποίος έχει αδιάκοπα αγωνιστεί για τις ελευθερίες και την ειρήνη. Αντίστοιχα πιέζονται η γυναίκα του, η συντροφή του και άλλες οργανώσεις ανθρωπιστικές. Ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολιτειών και άλλων αρχών έχει παγώσει από την σύλληψη και φυλάκισή του ο λόγο, η φυλάκιση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Ανεξαρτήτως της εθνότητας, της θρησκείας του, ο Λαντόχτη είναι ελεύθερος διανοητής που πιστεύει στην ειρηνική συμβίωση μεταξύ των διάφορων εθνοτικών ομάδων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Έχει επιμείνει για την ελευθερία της έκφρασης με όλες τις απειλές ε, της σύλληψης, της κατοίκων κράτησης, της φυλάκισης. Έχει καταγγείλει την ε, καταστολή εις βάρος και τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των Ουιγούρων αλλά και άλλων μειονότητων στην Κίνα. Έχει προσπαθήσει να συμβάλλει στο διάλογο ιδρύοντας ε, έναν ιστότοπο σε ουιγουρική και κινέζικη γλώσσα. Έχει μιλήσει για το γεγονός ότι είναι προετοιμασμένος και για μακροχρόνια φυλάκιση ακόμα και για θανατική ποινή εις του. Ελπίζοντας, λέει, ότι αυτό θα μπορούσε τουλάχιστον να συμβάλλει στην αφύπνιση για τα, τη σχετική με τα προβλήματα των Ουιγούρων. Πέρασε παράθεση. Αυτό επιδιώκει λοιπόν. Ναι, όχι πρόεδρε, τελειώνω. Έχει επιμείνει λοιπόν να καταγγέλει τις ε, διακρίσεις και τις πιέσεις βάρος του λαού των Ιγούρων με την ε, απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στον Ιλάν Τόχτη το Κοινοβούλιο θα αποστείλει ένα σαφές μήνυμα για το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, ανθρώπων και από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και θρησκευτικές πεπιθήσεις. Παρακαλώ τώρα και ευχαριστώ που σας με ακούσετε να δούμε το βίντεο.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 сөз пайдасыз сөз болған Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κανείς το λόγο για ερωτήσεις, για να υποστηρίξει κάποια υποψηφιότητα. Όλα είναι σαφή. Ωραία, τότε να σας εξηγήσω πώς θα προχωρήσουμε με το χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε ότι στις 11 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης, ΑΦΕΤ και ΔΕΔΕ. Η διάσκεψη των Πρόεδρων στη συνέχεια θα αποφασίσει για τον επικρατέστερο στις 27 Οκτωβρίου και στις 12 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, στο Στρασβούργο, θα γίνει συνεδρίαση πάλι κοινή όπου θα ανακοινωθεί ο βραβευτής και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι προβλέπεται η τελετή απονομής. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη βοήθειά σας και θα τα ξαναπούμε στις 11 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ.